ΕΛΚ έλαβα αιτήματα για διορισμούς και αλλαγές στις επιτροπές και ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται και μέχρι, αν δεν υπάρχει αντίρρηση μέχρι την έγκριση των πρακτικών θεωρούμε ότι εγκρίνονται αυτές.